Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's Foreign Affairs Committee. Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καλώ ορίσατε στη σημερινή συνεδρίαση. 8 λεπτά έχουμε αργήσει. Καλύτερα να ξεκινήσουμε. Ένα σύντομο μήνυμα από τι Γερμανίε. Βρισκόμαστε στη 36η ημέρα τη διαμαρτυρία μα κατά τη μονομερού επιβολή ε, όρων εργασία από πλευρά τη διοίκηση. Γι' αυτό η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώ την προβλεπόμενη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. αυτο η διερμηνια θα σταματησει ακριβω την προβληπομενη ωρα ληξη τη συνεδριαση ευχαριστουμε για την κατανόησή σα. Τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, μια και δεν έχω ανακοινώσεις, ε, ε έγκριση των ε, πρακτικών της 16ης Μαΐου, αν δεν έχετε αντιρρήσει θα εγκριθούν μέχρι το τέλος συνεδρίασης. Σημείο 4, ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Κάριν Κράισελ, ε, Υπουργό για την Ευρώπη, την Ολοκλήρωση και τις Εξωτερικές Υποθέσεις Αυστρίας, τρίτη φορά μετά το 1998 και 2006 που αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αυστρία συνοδεύεται από τον Αλεξάνδρ Μάρσικ, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας, τον μόνιμο εκπρόσωπο πρέσβη κύριο Νίκολας Μάρσικ, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή, α είναι, είναι εδώ, είναι συγγνώμη, δεν θα αργήσει, είναι εδώ ήδη, δεν τον είχα δει. Ε, εδώ στη σημειώση μου έχουν γράψει ότι μπορεί να καθυστερήσετε. Ποιο το γράψει αυτό. Κυρία Κνάισελ, είναι πολύ καλή συνήθεια στην αρχή της ε, κάθε προεδρίας να εμφανίζεται εδώ ο υπουργό εξωτερικών της προεδρεύουσας χώρας. Αυτή είναι η πιο καλή από τις επιτροπές της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έξι μήνες ε, πιο πριν είχαμε δει τον Βουλγαρό ε, Υπουργό Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της. Ε, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να παρουσιάσετε τις προτεραιότητες σας, προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας. Δεν υπάρχει διερμηνία προς τα Ολλανδικά σήμερα. Δεν βλέπω κανέναν Ολλανδό ή Φλαμανδό συνάδελφο έτσι κι αλλιώς. Ε, ε, Υπουργέ κυρία Κνάισελ, καλώς ήρθατε. Σα um, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε David McAllister. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα για άλλη μια φορά. Πριν ένα χρόνο περίπου είχα τη δυνατότητα να σας κάνω μια παρουσίαση εδώ σε τούτη την αίθουσα. Θα ήθελα να χαιρετήσω τα πρόσωπα που γνωρίζω. Βλέπω τον κύριο Πέτερλε, τον κύριο Φρόιντ και άλλους που έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Επανένωση, λοιπόν, είναι αγνωριμία για κάποιους άλλους από εσά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θέρμα τους διερμηνείς, λέει η κυρία Υπουργός, που θα διευκολύνει την επικοινωνία μας. Θα μιλήσω γαλλικά, μετά αγγλικά και μετά γερμανικά για να αναγνωρίσω την αρχή της πολυγλωσσίας. Αλλά βέβαια ε, ε, μπορείτε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας να μιλήσετε αγγλικά, τη lingua franca μας. Ε, θα κάνω και ό,τι μπορώ για να απαντήσω στα ισπανικά ή τα ιταλικά στο βαθμό που μπορώ. Είμαι ευγνώμων στους συναδέρφους που έχουν ετοιμάσει τη σημερινή μου ομιλία. Ξεκινώ λοιπόν στα γαλλικά, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα. Πρόεδρε, αγαπητέ Νταβίτ, αγαπητά μέλη, είναι τιμή μου και προνόμιο μου να απευθυνθώ σε εσά σήμερα ως Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας και ως ε, Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Παθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Είναι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στην νομοθετική διαδικασία, αλλά και ως ευρωπαϊκό όργανο που μεριμνά για, ε, για το διαχωρισμό των εξουσιών. Επί τη βάση αυτής της αρχής του διαχωρισμού των τριών εξουσιών έχει χτιστεί η Ευρώπη. Αυτή η αρχή αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και αυτή η αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών μας δίνει το χαρακτήρα που έχουμε. Τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αυτό που είπε ο Μοντεσκιό το 1748 που έγραφε στο πνεύμα των νόμων. Δεν υπάρχει ελευθερία αν η εξουσία η δικαστική εξουσία δεν είναι διαχωρισμένη από την εκτελεστική και την νομοθετική. Ο Μοντεσκιό εξακολουθεί να είναι ένας από τους αγαπημένους μου φιλοσόφους και, μας, και είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τις ε, βασικές αρχές οι οποίες μας δίδαξε εδώ και όχι τόσο πολύ χρόνο, τον διαχωρισμό των εξουσιών δηλαδή και το σεβασμό στο νομοθετικό έλεγχο. Είναι κάτι το οποίο σέβομαι από την αρχή της πολιτικής μου καριέρας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα. Αν, μου επιτρέπετε να συνεχίσω να αναφέρω τα λόγια του λέει, τα πάντα θα τα χάναμε αν ο ίδιος άνθρωπος ή το ίδιο όργανο ασκούσε και τις τρεις αυτές εξουσίες. Δηλαδή νομοθετούσε, εκτελούσε τις ε, αποφάσεις και δίκαζε ε, τις, ε, ε, τα αδικήματα. Τώρα αλλάζω στα, φέρουμε στα αγγλικά. Ε, αυτό θα, αυτή θα ήταν η, η, μόνη μου ε, επίσημη εμφάνιση εδώ πέρα, σύμφωνα με τη συνήθεια της αλλά θα ήθελα ε, να διοργανώσουμε ένα άτυπο διάλογο του επόμενους μήνες, ε, έτσι ώστε να ε, συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε τη συζήτησή μας. Αυτό ως μια συμβολική χειρονομία αυστριακής φιλοξενίας. θα σας... Ε, είστε οι πόρτες μου, η πόρτα του γραφείου μου θα είναι ανοιχτή αν βρεθείτε μάλιστα στη Βιέννη να φάμε μαζί ένα μεσημεριανό ή να με δείτε στο γραφείο μου. Για την Αυστρία αυτή είναι η πρώτη προεδρία μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, έχουμε διορίσει την κυρία Μογκερίνη, έχουμε αναθέσει το καθήκον να ηγηθεί της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αυστριακή Προεδρία στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ΥΠΑ της εκπροσώπου, της κυρίας Μογκερίνη. Και θα ήθελα να την ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τη Φεντερίκα και, την ομάδα της, του συμβούλου της, για το έργο της τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Φεντερίκα και ε, μου ήταν, εμφανίστηκε ξαφνικά μια σπίθα, ε, ένας ε, ξαφνικός έρωτας θα έλεγα, γιατί η εξωτερική πολιτική είναι για μένα το αντικείμενο της ζωής μου εδώ και πολλά χρόνια. Τους τελευταίους μήνες ξεκινήσαμε με μια πολύ καρποφόρα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και για να βελτιώσουμε την κατανομή των βαρών, το εννοώ, ε, πρέπει να προσπαθήσουμε ο καθένας μας να βάλει σε αυτό το κοινό τραπέζι τις ε, εμπειρίες του. Μπορούμε να αλληλοσυμπληρωθούμε. Κάποιες χώρες είναι πιο κοντά στην α περιοχή, κάποιες χώρες στη β, έχουμε διαφορετικές εμπειρίες και πρέπει να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Εγώ θα εκπροσωπήσω την κυρία Μογκερίνη όποτε χρειαστεί και θα προσπαθήσω να συνεργαστώ πολύ στενά μαζί της έτσι ώστε η εξωτερική μας παρουσία να είναι συνεπής. Πιο συγκεκριμένα η Αυστρία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυρίας Μογκερίνη προκειμένου να εφαρμοστεί η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα πάρουμε τη σκητάλη και της Βουλγαρίας και της Εστονίας καθώς σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε το τρίο των Προεδριών. Όπως γνωρίζετε, έχουμε συμφωνήσει ένα πρόγραμμα 18 μηνών εστιασμένο στα τέσσερα εξιστέματα. Πρώτον, μια ένωση την απασχόληση. Δεν μιλώ για δουλειές. Άλλο δουλειά, άλλο απασχόληση. Το κάνω ε, σκοπίμως. Να μην αναφέρομαι σε θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε απασχόληση εκεί που ο καθένας είναι προετοιμασμένο στον τομέα που είναι προετοιμασμένο. Δεύτερον, μια ένωση που θα ε, προστατεύει τους πολίτες, όλους τους πολίτες, με μια πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική που θα είναι σταμένη στο μέλλον, με μια πολιτική δικαιοσύνης και ασφάλειας ικανοποιητική που θα καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο παίκτη περαιτέρω η Αυστριακή Προεδρία θα εργαστεί σε ένα μεγάλο αριθμό περίπλοκων ζητημάτων που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Εσωτερική εξωτερική ασφάλεια, προστασία των εξωτερικών συνόρων, μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματο ασύλου, διεύρυνση τη πολιτική ε, γειτονία και ε, συμπλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον Brexit, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Τέλο, ποιε είναι οι δικέ μα προτεραιότητε. Η, το πρόγραμμα της Αυστριακής Προεδρίας που έχει ως ε, σύνθημα Ευρώπη προστατεύει ε, θέλει να δώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να απαντάει στις ανάγκες των πολιτών αμέσως όταν μόλις παρουσιάζονται. Θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φτάσει πιο κοντά στους πολίτες της και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους. Γιατί έχουμε χάσει τους πολίτες μας. Κάποια στιγμή στο δρόμο σε ορισμένε χώρε. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στη δράση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς θα πρέπει να είναι μια δύναμη σταθερότητας και σταθεροποίηση στον κόσμο. Η Αυστριακή Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη που προστατεύει. Και να σας πω ποιε είναι οι τρεις προτεραιότητες σε αυτό το θέμα. Πρώτον, Ασφάλεια και μετανάστευση. Δεύτερον, διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της χρήσης τεχνολογίας. Η λέξη κλειδί είναι ρομποτική, είναι ψηφιοποίηση, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ δείχνει να χάνουμε τεχνολογικό πεδίο έναντι χωρών στην, όπως για παράδειγμα στην ε, Ανατολική Ασία. Ε, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το πόσο σημαντικό και επίγον είναι αυτό ε, να πληρωθεί το αυτό το κενό. Τρίτον, σταθερότητα στη γειτονία με περαιτέρω προσέγγιση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Δυτικών Βαλκανίων, όταν, για όσοι από με γνωρίζουν ή έχουν ακούσει συνεντεύξεις μου, Προτιμώ να μιλώ για την Ανατολική Ευρώπη και όχι για Δυτικά Βαλκάνια. Δυτικά Βαλκάνια είναι τεχνητό. Σεράγεβο, Βελιγράδι, Σκόπια και άλλε είναι ευρωπαϊκέ πόλει. Όποιο έχει πάει στη φυλα... στην αίθουσα τη φιλαρμονική του Σεράγεβο ή στην ε, Εθνική Πινακοθήκη του Βελιγραδίου ξέρει ότι αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης και όχι ε, κάποιας, κάποιου αόριστου δημιουργήματος φαντασίας. Τώρα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Είναι σημαντικό να εργαστούμε πιο στενά με τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίσουμε την, την αποτελεσματική λειτουργία των πολιτικών επιστροφών. Ο διάλογος για θέματα μετανάστευσης θα πρέπει να εστιαστεί σε συγκεκριμένες χώρες προέλευσης ε, σύμφωνα και με το μοντέλο των υπαρχουσών ε, συμφωνιών σύνδεσης και εταιρικής ε, σχέσεις. Για παράδειγμα, χώρες της Βόρειας Αφρικής, ε, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη δημογραφικές αλλαγές, να δημιουργηθούν στενές εταιρικές σχέσεις με τις αφρικανικές χώρες που θα, θα, ε, θα εκπληρώσει τι ανάγκε και τι επιθυμίε και των δύο πλευρών. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ στο παρελθόν. Η Αυστριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στη σύνδεση με την ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν τρίτες χώρες που θέλουν να συνεργαστούν στην επανεισδοχή ε, πολιτών τους. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε δει αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας εις βάρος της αναπτυξιακής βοήθειας. Θα μιλήσω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό αύριο. Είναι επίση σημαντικό να δίδουμε συνδρομή σε όσου χρειάζονται προστασία πριν εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά είναι σημαντικό να προλάβουμε την είσοδο αυτών που δεν χρειάζονται ε, διεθνούς προστασίας. Οι αρχικοί κρατών κυβερνήσεων θα συζητήσουν αυτά τα θέματα στην άτυπη διάσκεψη κορυφή στο Σαλτσβούργο στι 20 Σεπτεμβρίου και θα δώσουν συνέχεια στην μεταναστευτική ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την ε, κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας, ε, επιθυμούμε είπατε εκπρόσωπο εκπρόσωπος να υλοποιήσει την παγκόσμια στρατηγική μας με προτεραιότητα στα εξή. Αύξηση τη ασφάλεια και τη σταθερότητα στην άμεση γειτονιά μα, προωθώντα την ευρωπαϊκή προοπτική στην νοτιοανατολική Ευρώπη, προωθώντα ε, μια διεθνή τάξη βασίζεται σε κανόνε και ενισχύοντα τι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασία. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ε, έθεσα ως προτεραιότητα την Ασία, γιατί το τελευταίο βιβλίο που είχα δημοσιεύσει ήταν «Αλλαγή φρουράς κινούμενοι από ένα, μια παγκόσμια τάξη που διέπεται ε, αντί από τις Πολιτείες, από τη σχέση, από τη σχέση με την Ασία. Σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και για την οικονομία και για στρατηγικούς λόγους. Θα σας δώσω ίσως περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, να σας πω όμως τις βασικές ε, αρχές γι' αυτό. Αναγνωρίζω πολύ καλά ότι φύσταται κάποιο σκεπτικισμός. Όμως, αυτό που μας λείπει, νομίζω, είναι γεωπολιτική σκέψη, πραγματική αυθεντική γεωπολιτική σκέψη. Πολύ συχνά απασχολούμαστε πιο πολύ με τα καθημερινά, με την καθημερινή διαχείριση, τα, τα μικρά και περιορισμένα, αντί να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο. κυρία είναι εδώ, μόλις έφτασε, και ε, έχοντας ε, σπουδάσει στη Γαλλία μπορώ να πω ότι μοιήθηκα στην γεωπολιτική σκέψη. Και αυτό θα πρέπει να το ενισχύσουμε, να το ενισχύσουμε και στη δική μας δουλειά. Οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Δεν μπορεί κανείς να τις αγνοήσει. Αλλά δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε σε αυτές. Πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Η νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί να κινδυνεύσει να πέσει σε κάποιο είδου κενό, το οποίο θα πληρώσουν, θα συμπληρώσουν πολύ εύκολα κάποιοι άλλοι. Ή γιατί ενδεχομένω θα προσφέρουν καλύτερε τιμέ. Μιλώντα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο στόχο τη Προεδρία μα είναι να ενθαρρύνουμε του εταίρου μα, όπω για παράδειγμα τη Βόρεια Μακεδονία, την πρώην Φύρομ, να ακολουθήσει το δρόμο της ένταξης. Θέλουμε να συνεχίσουμε διαπραγματεύσεις γρήγορα με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, όπως ακριβώς το ανέφεραν και τα συμπεράσματα της 26 Ιουνίου. Ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και τις προκαταρκτικές εργασίες για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε θέματα που είναι σημαντικά και για τις δύο πλευρές, την περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο οι εταίροι μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη θα συμμετάσχουν σε επιλεγμένες συζητήσεις που θα γίνονται μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, δύο χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υποψήφιες και ενδεχόμενες υποψήφιες, και η Τουρκία, συγγνώμη, έξι εταίροι από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Τουρκία, θα προσκληθούν σε ένα γεύμα εργασία μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, το Κίμλιχ, στι 31 ε, Αυγούστου μαζί με τους συναδέλφους τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντο. Επιπλέον, η Αυστρία θα συνεργαστεί στενά με τις χώρες περιοχής για πολύ συγκεκριμένα θέματα όπως για παράδειγμα την επίλυση διμερών διαφορών κατόπιν Τη Συνόδου τη Βιέννη τη διαδικασίες του Βερολίνου του 2015. Και υπάρχουν καλέ ειδήσει από αυτήν την περιοχή. Μπορούν αυτές οι, αυτές οι ειδήσει να δράσουν ως ενθάρρυνση. Ασφαλώς θα πρέπει να περιμένουμε τα δημοψηφίσματα, αλλά θα θέλω να συγχαρώ τους διαπραγματεύς, για, διαπραγματευτές ε, της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας για την επιμονή τους και την υπομονή τους. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Εγώ ποτέ δεν θα γινόμουν καλή διπλωμάτηση, πολύ καλή διπλωμάτιση, γιατί μου λείπει η υπομονή. Αλλά ε, θέλω να ποτίσω φόρο τιμής στο κουράγιο τους, στη γενναιότητά τους. Χρειάζεται γενναιότητα γι' αυτό που έκαναν. Ε, αποτελεσματική πολυμέρεια. Τι σημαίνει αυτό. την ε, πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, GCPOA. Γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, το Μάιο αποσύρθηκαν από αυτή τη συμφωνία. Βρισκόμαστε σε ένα λίμπο. Οι Ιρανοί προσπαθούν να ε, ζητούν τη βοήθειά μα για να σώσουμε τη συμφωνία. Το έχω πει και στο παρελθόν. Να σα πω ποια είναι η δική μου πεποίθηση. Ο κίνδυνος δεν είναι απλώς να χάσουμε μια συμφωνία αφοπλισμού. Η απειλή είναι να χάσουμε την αξιοπιστία μας. Και όταν μιλούμε για αποτελεσματική πολυμέρεια και μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, αυτό το λέει κάποιο ο οποίος δίδασκε διεθνές δίκαιο, έτσι. Και γνωρίζω ότι το διεθνές δίκαιο υποφέρει τουλάχιστον από τον πόλεμο του Ιράκ και μετά. Όμως η αξιοπιστία δεν αγοράζεται στο σούπερ μάρκετ, κερδίζεται. Και με την συμφωνία του Ιράν, αυτό που διακυβεύεται είναι αυτό ακριβώς η αξιοπιστία. Και εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μαζί με την ομάδα της Φεντερίκα Μογκερίνη. Και με τα άλλα συμβαλόμενα μέρη της ε, συνθήκης. Τώρα, ρόλος μας ως χώρα που φιλοξενεί διάφορα όργανα του ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ, Οργανισμό ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. Ω ε, τέτοια χώρα ε, έχουμε ανάγκη να διατηρούμε το διάλογο και να ε, τον συντηρούμε. Τώρα, εμβάθυνση το σχέσεων με την Ασία, επανέρχομαι. Η νέα στρατηγία, ευρωπαϊκή στρατηγία τη σύνδεση με την Ασία θα είναι η βάση για την οικοδόμηση πιο στενών δεσμών μεταξύ των δύο περιφερειών. Η σύνοδος κορυφής που θα οργανώσουμε θα είναι το πιο σημαντικό γεγονός η κορονίδα. Οι εξωματούχοι ήδη συναντήθηκαν στη Βιέννη την περασμένη εβδομάδα και οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΑΣΕΑΝ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα συνεργαστούν να συζητήσουν τη συνεργασία μα. Όπω πάντα στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ο Νίκολα Τάλεπ ε, είχε γράψει το 2008 το βιβλίο το, το «Μαύρη κύκνη» ε, για, ακριβώς για τα πρόβλεπτα γεγονότα τα οποία μπορούν να αλλάξουν το ορμό της ιστορίας γεγονότα τα οποία όμως έχουν συγκεκριμένους, συγκεκριμένες αιτίες, αίτια. Και θα πρέπει λιγάκι να το σκεφτούμε. Θα ήθελα να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους γεγονότα. Μας ανισχύει ιδιαίτερος η κατάσταση στην Ιεμένη, στην Λωρίδα της Γάζας και γενικότερα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τις διπλωματικές προσπάθειες που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν κάτι που να μοιάζει με ασφάλεια και ειρήνευση και συμφιλίωση. Συνεργασία με τις ε, πολιτείες και, το, και διατλαντικός διάλογος. Γνωρίζουμε ότι τα όσα θα συμβούν, τα όσα συμβαίνουν σήμερα εδώ ε, μπορεί να αφήσουν σφραγίδα, αλλά περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Καλωσορίζουμε ε, τα συμπεράσματα για τη συμφωνία μετά το Κοτονού. Προετοιμαζόμαστε για την υπουργική συνεδρίαση με τις ε, χώρες Λατινικής Αμερικής, της ΣΕΛΕΚ, είναι η εταίροι μα ε, για τη νέα στρατηγική Ελληνική Αμερική κατά τη διάρκεια Προεδρία μα. Τελειώνοντα, αναφέρουμε στην εφαρμογή τη παγκόσμια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασφάλεια. Για να προβάλλουμε τι φιλοδοξίε μα. Χρειάζεται να συνεργαστούμε με πολυμερή οργανώ όπω ο ΙΕ, το ΝΑΤΟ, ε, η Αφρικανική Ένωση και ο ΑΣΕ οι διμερείς δράσεις εξακολουθούν να δεσπόζουν, αλλά δικό μας καθήκον είναι να θέσουμε ε, εμπόδια στην άνοδο αυτής της τάσης για διμερείς πρωτοβουλίες. Καταλαβαίνουμε βέβαια τις ανησυχίες των πολιτών σε ό,τι αφορά, αφορά, για παράδειγμα, την παγκοσμιοποίηση. Οπότε δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει αυτό που συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να το δαμάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αναμένω να συνεργαστούμε με όλες τις μόρφες που μπορούμε, χωρίς το δικό σας νομοθετικό έλεγχο των δικών μας δράσεων, η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ κυρία Κνάλης για την επισκόπηση του προγράμματος ε, της Αυστριακής Προεδρίας. Συνήθως το κάνουμε ως εξή. Οι συνάδελφοι θέτουν ερωτήσεις ε, και στο τέλος θα μπορέσετε να συνοψίσετε με ενημέρωσαν ότι πρέπει να φύγετε ακριβώς την ώρα σας. Έχουμε δηλαδή ακόμη 25 λεπτά μέχρι τις 3.30. Αυτή τη στιγμή 8 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. 10. Παρακαλώ να περιοριστείτε στο 1-1,5 λεπτό. Ξέρω ότι είναι φιλόδοξο αυτό, αλλά ας προσπαθήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τον Κρίστιαν Πρέντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και να παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Εγώ θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει σχέση με αυτό που ονομάζετε εσείς Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εμείς ε, συνήθως μιλάμε για Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη γνώμη σας για τη Βοσνία Αργαζεγοβίνη, μιας και το φθινόπωρο θα γίνουν εκλογές και επίσης δεδομένης της μεταναστευτικής κρίσης. Έτσι εκλαμβάνεται πάντως στην Βοσνία Αργαζεγοβίνη. Και φαίνεται οι αρχές εκεί είναι λίγο χαμένες. Δεύτερη ερώτηση. Το... Συζητήσαμε το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια ή Μολδαβία. Στα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ζητήσαμε να μην ε, σταλεί κανένα ευρώ πριν αποκατασταθεί η λειτουργία της δημοκρατίας. Εσείς πότε το βλέπετε η κατάσταση στη Μολδαβία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλέκενστάιν. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που μόλις είπε ο Κρίστιαν Πρέντα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Με πολύ χαρά άκουσα, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς και οι συνεργάτες σας παρουσιάσατε ακριβώς αυτήν την οδό πριν από μία εβδομάδα ε, στο Συμβούλιο πολύ προσεκτικά, ίσως υπερβολικά προσεκτικά. Τονίσατε την ανάγκη για σταθερότητα. Αναφερθήκατε στην μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στην Αλβανία και σε άλλα θέματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι θέμα αξιοπιστίας να παρουσιάσουμε αποτελέσματα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στηρίξετε τους φίλους μας ε, στην Μακεδονία, λέει ο μιλητής. Ε, δημοψήφισμα τους περιμένει και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι χαιρόμαστε πολύ που βρήκανε μία λύση μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και ίσως θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο ο Ομοσπονδιακός ε, Καγκελάριος να συμμετάσχει στην προσπάθεια. Νομίζω ότι αποτελεί πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε ποια είναι η θέση μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φλέκενστάιν, ο Τσάρλ Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Κνάισλ, ήταν ε, εξαιρετική επισκόπηση που μας δώσατε. Εμένα με ανησυχεί πολύ το θέμα του αποτελεσματικού της ε, αποτελεσματικής πολυμερούς μεθόδου. Υπάρχει μια ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα την οποία θα πρέπει να προσέξουμε. Ιδιαίτερα με ανησύχησε το θέμα της πολυμέρειας όταν άκουσα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτών να λέει ότι πιο πολύ τον απασχολούσε η συνάντησή του με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και την κυρία Μέη παρά η συνάντησή του με τον πρόεδρο Πούτιν. Εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργη αυτή η δήλωση από πλευράς του ηγέτη του ελεύθερου κόσμου. Ε, και φοβάμαι κιόλας ότι αν τον αφήσουν μόνο του με τον Πούτιν θα προσπαθήσει να επαναχαράξει τους χάρτες στην Δυτική Ευρώπη και ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, σε λίγο θα συζητήσουμε την έκθεσή μου για το Μαυροβούνιο. Και Σκεφτείτε το θέμα της Ουγγαρίας, ε, της Ουκρανίας, ε, σκεφτείτε τι θα γίνει αν ξαφνικά ο Πούτιν μαζί με τον Τραμπ ε, δηλώσουν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αναγνωρίσουν την προσάρτηση της Ουκρανίας ή την απόσχηση της Τραμπας ή άλλων περιοχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ εύκολες ερωτήσεις. Ήβο Βάιγκλ από την Άλντε, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω στο Κοινοβούλιο. Πολύ χαίρομαι που ως πρώην δημοσιογράφος έχετε καταρτήσει ένα πολύ πλήρες πρόγραμμα. Διακρίνω το πνεύμα της ελεύθερης σκέψης στο πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Ε, και επίσης έχετε αναλάβει τα ενία μιας εξαιρετικής διπλωματίας. Δεν έχω τίποτα να πω για τις προτεραιότητές σας, πάρα πολύ καλά δομημένες είναι. Θα ήθελα μόνο να σας ρωτήσω το εξής και θα θέσω στα, στα σλοβένικα την ερώτησή μου για να ακουστεί άλλη μια γλώσσα. Ευρώπα. Ευρώπη... Ε, Η Ευρώπη φαίνεται να βρίσκεται σε μια, εν μέσω μιας πολιτικής μετάβασης και μας ανησυχεί πολύ. Ανησυχούμε ότι τελικά δεσπόζει η λογική του λαϊκισμού, του εκφοβισμού και της ξενοφοβίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό ως πολιτικός από την Αυστρία. Πώς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν θέλουμε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μια φτηνή πολιτική που να βασίζεται στον λαϊκισμό και ε, τον λαϊκισμό. Ευχαριστώ κύριε Βάγκελ. Η Ρεμπέκα Χάρμς. Κυρία Υπουργέ, εμένα με ενόχλησε που δεν είπατε τίποτα για την πολιτική γειτονία και την Ανατολική Ευρώπη, διότι η Αυστρία συχνά έχει επικρίνει αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τσάλς Τάνοκ σας έθεσε μία ερώτηση. Θα ήθελα και εγώ να γνωρίζω πώς θα διαμορφώσει στη συνέχεια η Αυστρία την πολιτική αυτή. ο ΑΣΕ, το θέμα του Ντάμπας. Είχαμε εδώ έναν ομιλητή πριν δύο εβδομάδες που είπε ότι οι δύο τελευταίοι μήνες ήταν οι πιο αιματηροί. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει τι θέλουν να κάνουν εκεί οι Αυστριακοί. Επίσης, έχουμε εδώ μια οξία κρίση. Η Ρωσία στην ε, Αζωφική θάλασσα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Βλέπουμε μία κλιμάκωση η οποία όμως ε, κρύβεται αυτή τη στιγμή πίσω από το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ, Ρεβέκα Χάρμς. Thank Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο μίλησε ε, πρέπει να διαπιστώσουμε πώς θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και να αναλύσουμε την ε, πρόσφατη απόφαση για αυτό το θέμα. Καταρχήν σε ό,τι αφορά το Brexit, δεν νομίζω ότι είπατε και πολλά πράγματα. Βασικά δεν είπατε τίποτα. Θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεύτερον, συμφωνείτε ότι η Ευρώπη υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί εξαιτία όλων αυτών των προβλημάτων. Thank you. And now for the, the EFTD group is... Ευχαριστώ. Για το ονόματο τη ΕΝΕΦ, η κυρία Ορκέσιο. Καλωσορίζω την Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας που ε, έκανε μια πλήρη ε, ε, παρουσίαση της κατάστασης διεθνές επίπεδο και των θεμάτων που απασχολούν τις κυβερνήσεις. Και τι, θα γίνει, τι σκοπεύει να κάνει η Αυστρία για να ε, διαχειριστεί το πρόβλημα της, ε, της διακίνησης ε, ανθρώπων, της εμπορίας ανθρώπων, κάτι που επηρεάζει πολύ αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερθήκατε συγκεκριμένα στην αποτροπή των αποχωρήσεων. Εμένα η ερώτησή μου είναι εξής. Ποιες πρωτοβουλίες ε, θα ληφθούν ε, κατά διάρκεια της Αυστριακής ε, Προεδρίας για να έχουμε μια μεγαλύτερη επιρροή, γιατί Μιλήσατε για την πολιτική δράση της ε, κυρίας Μογκερίνη με εξαιρετικά λόγια, αλλά τα αποτελέσματα είναι λίγα σε αυτό το τομέα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να έχετε κάποια επιρροή. Συμφωνείτε επίσης με αυτό που είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά που δεν έλαβε στήριξη από την Κομισιόν Δηλαδή την όθηση να δημιουργηθεί ένα ε, σχέδιο Marshall για την Αφρική, γιατί από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ πιθανό. Ευχαριστώ πολύ. Ο James Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η αδύναμη νόμη είναι άχρηστη νόμη. Εμένα η ερώτησή μου αφορά την Γεμένη, μιας και αναφερθήκατε στην συμφωνία με το Ιράν. Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει ε, πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και τη Συμμαχία ή πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανή μια εσωτερική σύγκρουση. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, James Carvin. Έχουμε ομιλητή από κάθε πολιτική ομάδα. και ο κύριος Μέζεριτ, ξέχασα να τον αναφέρω. Ε, συμφωνήσαμε ότι θα μείνετε 10 λεπτά περισσότερο, έτσι δεν είναι. Ωραία. Παρακαλώ. Κυρία Υπουργέ, καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπατε ότι προτιμάτε την, τον όρο Νότιο-Ανατολική Ευρώπη για να περιγράψετε την, το, τη συνολική περιφέρεια. Ένα από τα προβλήματα της στρατηγικής ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ότι ε, πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπαίδιο. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα Σερβίας-Κωσυφοπεδίου και αυτό συνδέεται με την πρωτοβουλία της Κομισιόν ε, του Σεπτεμβρίου ή του Οκτωβρίου ε, στην εξωτερική πολιτική να περάσουμε από την ομοφωνία στην ε, πλειοψηφία πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις δράσεις μας. Σε συνέλευση του ΟΗΕ το βασικό μήνυμα θα πρέπει να είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με ενωμένη φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος αυστριακός συνάδελφος, ο κύριος Φρόιντ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να πω αυτό που είπα και στον Καγκελάριο στο Στρασβούργο. Ευχόμαστε επιτυχία στην Προεδρία σας. Ε, υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Ένα σχετίζεται με το θεματολόγιο σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμπίπτει στη δική σας αρμοδιότητα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί και τι σημαίνει αυτό για σας. Και δεύτερον, που μπορεί να μην ε, είναι ακριβώ θέμα ενόχληση, αλλά υπάρχει μια γενική ευρωπαϊκή ενόχληση, είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη σχέση αυτή. Και τρίτον, το δικό μου σύνθημα, το δικό μου μάντρα. Για να έχουμε ενωμένη και συνειδητή εξωτερική πολιτική. Συμφωνείτε να ξεφύγουμε από την αρχή της ομοφωνίας στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Το μας Μέζοριτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, για την παρουσίασή σας. Ήταν πράγματι πολύ ευρία και προχώρησε και εις βάθος ταυτόχρονα. Ε, τι έχετε μπροστά σας στο, στο πιάτο σας, για να το πούμε έτσι το Κοινοβούλιο έχει διαμορφώσει τη θέση του σχετικά με έναν ε, μελλοντικό κανονισμό του Δουβλίνου. Το Συμβούλιο που βρίσκεται στο θέμα αυτό. Και δεύτερον, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι ο μικρός κυβερνητικός εταίρος δεν θα επηρεάσει την πολιτική της κυβέρνησής σας και της Προεδρίας σας όσον αφορά τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τέμας. Ο κύριος Πέτερλε. Πολύ χάρηκα που άκουσα τις φιλοδοξίες της Αυστριακής Προεδρίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Και χαίρομαι πολύ που σας ενδιαφέρει η συνεκτικότητα στις εξωτερικές πολιτικές. Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, έχουν τεθεί πολλές ερωτήσεις. Η δική μου ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Αναφερθήκατε και στην Ασία. Πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις της σχέσης μας με τη Ιαπωνία, διότι δύο σημαντικές συμφωνίες θα υπογραφούν αύριο για την ε, στρατηγική και επενδυτική εταιρική σχέση. Πώς θα επηρεάσει αυτό τη σχέση στο μέλλον. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το προσέχες εξάμεινο. Ευχαριστώ. Alois Peterle, and finally our friend Milan Mon. Και ο φίλος μας ε, Φιλαν Μόν. Καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ. Θέλω να αναφερθώ στην ε, συνάντηση με την ΘΕΛΑΚ, την ε, συνάντηση με τους υπουργούς των χρόνων της Αντίνικης Αμερικής. Έχουμε τα προβλήματα της Βενεζουέλας και της Νικαράγουας. Γνωρίζετε τα, τη θέση του Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα. Πρόσφατα ψηφίσαμε και για τη Βολιβία και, πριν από δύο μήνες για την, για, και για τη Βενεζουέλα και πριν από δύο μήνες για την Νικαράγουα. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσετε το θέμα της συμφωνίας με τις χώρες του Μερκοσούρ. Θα μπορούσατε να μας ε, πείτε μερικά πράγματα παραπάνω για τις προθέσεις σας. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε ένα θέμα. Η διάσκεψη κορυφή των Δυτικών Βαλκανίων πραγματοποιήθηκε χθε και σήμερα και εσεί η ίδια είπατε ότι θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καθότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε προσέξει ιδιαίτερα το θέμα της Αλβανίας και της Μακεδονίας, θα θέλαμε η Αυστρία στο δεύτερο εξάμεινο να, να παίξει σημαντικό ρόλο. Οι δύο αυτές χώρες, εάν σημειώσουν πρόοδο στο δεύτερο εξάμεινο, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε νέα κεφάλαια. Η Αυστρία παραδοσιακά έχει πολύ στενέ σχέσεις με τις χώρες αυτές. Ελπίζουμε λοιπόν να παίξετε επικοδομητικό ρόλο και να μπορέσετε να στηρίξετε τις χώρες αυτές. Στο μεταξύ, είπατε ότι μπορείτε να μείνετε 10 λεπτά παραπάνω. Έχετε λοιπόν 16 λεπτά συνολικά για να απαντήσετε ε, στα πολλά αυτά θέματα για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Την ερώτησή σας να τη συνδυάσω αυτήν του Ρουμάνου συναδέρφου. Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Μολδαβία. Τον Οκτώβριο, μετά τις εκλογές, σκοπεύω να μεταβώ στο Σαράγεβο και τον τον Φεβρουάριο ε, στο Σαράγεβο είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Μου είπαν ότι θα πρέπει να μας βοηθήσετε και εγώ είπα ότι η βοήθεια δεν είναι αποτελεί διπλωματική κατηγορία. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ε, τα συμφέροντα που συγκλίνουν και πιστεύουμε ότι συμφέρει, είναι προς συμφέρον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης όχι μόνο να ε, αναθεωρήσει τον εκλογικό νόμο, αλλά να βελτιώσει και το επίπεδο ασφαλείας στη χώρα. Όσον αφορά τη Μολδαβία, γνωρίζω τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσωπικά θα ασχοληθώ με το θέμα. Την επόμενη εβδομάδα θα μεταβώ στο Βουκουρέστι και στο Τίσναο Θα ήθελα όμως πρώτα να συνεννοηθώ με τους αδέρφους μας και την Φεντερίκα Μογκερίνη ε, για να ακολουθήσω την κατεύθυνση των ε, δικών τους ψηφισμάτων. Ο συνάδελφος Μακάλιστερα αναφέρθηκε και στην πρόοδο που απαιτείται. Ναι, θα πρέπει πάντα να ε, αμείβουμε τα καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί. Στο Βελιγράδι είδαμε απελευθέρωση των θεωρήσεων. Κάποια τέτοια μέτρα τα βλέπουμε με σκεπτικισμό. Η σερβική πολιτική απελευθέρωση ε, από τις θεωρήσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται να ακολουθεί την ευρωπαϊκή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μεγάλο μέρος της λαθρομετανάστευσης πραγματοποιείται μέσω Βελιγραδίου. Πρέπει λοιπόν να πληρούνται κριτήρια και οι παροχές ε, να ακολουθούν τα καλά αποτελέσματα από πλευράς των χωρών αυτών. Κύριε Φλέκενστάιν, Αναφερθήκατε στην Βόρεια Μακεδονία, να την ονομάσω έτσι, αυτό θα είναι το μελλοντικό όνομα. Τα Σκόπια, είπατε ότι πρέπει να στηρίξουμε τα Σκόπια. Το τελευταίο εφτάμινο έχω πολύ ε, καλή επαφή με τον ε, εξω, ε, Υπουργό Εξωτερικών ε, Δήμητροφ και τον κύριο Κοντζιά και νομίζω ότι οι δύο αυτοί υπουργοί συνεννώνται πολύ καλά μεταξύ τους ε, και ε, θα έχω τη δυνατότητα να τους καλωσορίσω και εγώ. Πάντως εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε το θάρρος αυτών ε, των δύο ανθρώπων να αποφέρει καρπούς. Εσείς με ρωτήσατε σχετικά με την ευρύτερη εικόνα των Τραμπ και των Πούτιν. Ενώ θέτατε αυτή την ερώτηση, εμένα μου ήρθε μια παλιά εικόνα στο μυαλό από μια διάσκεψη πριν πολλά χρόνια. Έχω διαβάσει πολλά κείμενα του Winston Churchill που για μένα ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε την αυταπάτη των στενών σχέσεων. Δηλαδή αυταπάτη ότι αν δύο άνθρωποι τα πάνε καλά μεταξύ τους όλα είναι καλά. Όχι, υπάρχουν εθνικά συμφέροντα. Και θα μπορούσα να απαντήσω ως εξή στην ερώτησή σας. Πριν κάποιες εβδομάδες είδα έναν Ισραηλινό ε, συνάδελφο, είναι πολιτικός αναλυτής και ήρθε στο γραφείο μου, περιγράφοντας τον πρόεδρο Τραμπ ως εξή. Έχει ένστικτο, όχι όμως στρατηγική. το περιβάλλον του, θα πρέπει να το χειριστεί αυτό με κάποιο τρόπο. Στις μέρες μας, μας λείπουν άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουν ποια είναι τα συμφέροντα και να μην επισκιάζεται αυτό το επίκεντρο από τη χημεία μεταξύ ανθρώπων που μπορεί να βοηθάει αλλά δεν αποτελεί την αυτόματη λύση για τα πάντα. Να παραθέσω τα λόγια του Λόι George που το 1919 είπε ότι τι χρειαζόμαστε τους διπλωμάτες είναι σπατάλη χρόνου και χρημάτων. Και η Μάργαρετ Μίλαν στο βιβλίο της αναφέρεται στις συνθήκες του έτους αυτού, του 1919. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος, αλλά ας εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που χειρίζονται τα θέματα αυτά. Μερικές φορές οι διπλωμάτες, τα πρωτόκολλα εξυπηρετούν κάποιον καλό σκοπό. Ιβο Βάιγκλ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Μετά από τόσα χρόνια. Θυμάμαι τις συνομιλίες μας ε, τότε που ήμουν ε, διπλωμάτης ε, στην Σλοβενία και στην Λουμπλιάνα και σε πολλές άλλες ωραίες πόλεις της Σλοβενίας συναντηθήκαμε και η ερώτησή σας ήταν για την ξενοφοβία και τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό. Πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτές τις φτηνές μορφές πολιτικής. Θα πρέπει να οξύνουμε το κριτικό πνεύμα. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Θα ήθελα όμως να πω επίσης Και εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο λαϊκισμός. Το πρόβλημα που θα πρέπει να λύσουμε είναι μάλλον επιθυμίες, νοσταλγίες, φόβοι που υπάρχουν. Ε, στην, εισαγωγική μου ομιλία είπα ότι πρέπει να να, ε, να ξαναβρούμε την επικοινωνία με τους πολίτες. Και αυτό είναι το θέμα. Προσπαθώ να είμαι ρεαλίστρια. Να φροντίσουμε να μην μας στριμώξουν σε καμία αγωνία, να ε, προσανατολιζόμαστε πάντα με βάση την πραγματικότητα. Ρεμπέκα Χάρμς. Ε, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Ε, στην Φραγκφούρτη, στον Όντερ, είχαμε συναντηθεί το 2011, νομίζω, σε μια συνάντηση για την ενεργειακή πολιτική. Η μομφή σας είναι σωστή. Ε, δεν ε, είχα πολύ χρόνο για την ομιλία μου και γι' αυτό παρέλειψα κάποιε παραγράφου. Αλλά ναι, αναφερθήκατε στην ε, Ουκρανία και την Ανατολική Ουκρανία. Δεν έχω βρεθεί ποτέ στην Ανατολική Ουκρανία. Πέρασα όμως τρεις μέρες στην Δυτική Ουκρανία. εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε όλο αυτό το θέμα είναι πώς μπορούμε στην Ανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια Ντόνπας, να ε, δώσουμε ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης στους ανθρώπους εκεί. Έχουμε ειδικό εκπρόσωπο στην περιφέρεια αυτή, τον πρέσβη Μάρτιν Σάιντεκ, που ασχολείται με την ε, συνεργασία στην περιφέρεια αυτή και έχουμε διπλωμάτες που ε, εφαρμόζουν την πραγματική διπλωματία, προληπτική διπλωματία που κανείς δεν γνωρίζει ότι πραγματοποιείται. Κανείς ε, δεν παίρνει βραβείο θάρρους παράσημο για την προληπτική διπλωματία. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντική δουλειά αυτή. και με τους Ρώσους και με τους Ουκρανούς συναδέρφους είχα επανειλημμένα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και αυτό που με απασχολεί εμένα είναι η καθημερινή ζωή των ανθρώπων εκεί πώς είναι. Και άλλωστε δεν φταίει ποτέ μόνο η μία πλευρά. Σας ευχαριστώ όμως πολύ για την ερώτησή σας. Είναι ένα θέμα που παρέλειψα να αναφέρω κατά την εισαγωγική μου ομιλία. Η επόμενη ερώτηση ήταν του κυρίου Χατζηγεωργίου. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ είναι ο αρμόδιος διαπραγματευτής. Είχα δύο συναντήσεις μαζί του. Το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει τον Οκτώβριο. Ήδη τον Φεβρουάριο σχεδίασα μετάβαση στην ε, Ιρλανδία και γνωρίζουμε ότι το θέμα της Ιρλανδίας είναι πολύ σημαντικό στις διαπραγματεύσεις του Brexit, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, διότι πρώτον ο ε, διαπραγματευτής είναι ο κύριος Παρνιέ και δεύτερον αλλάζουν τα πράγματα ώρα με την ώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέθηκε η ερώτηση, μπορεί να διαλυθεί η Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε περάσει πιο δύσκολους καιρούς. Θυμάμαι την άνοιξη του 2003 που ακούσαμε διάφορες δηλώσεις πριν, ε, για τον επικείμενο τότε πόλεμο στο Ιράκ. Ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θυμάμαι ότι είχε πει δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Υπήρχαν διαφωνίες, διαμάχες σε πολλούς τομείς. Ναι, και σήμερα έχουμε χάσματα, Έχουμε ε, τις διαφορές βορρά-νότου, ανατολής και δύσης. Αλλά ας αφήσουμε την Ευρώπη να ενεργήσει εκεί που μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα και να μην ε, σπαταλάμε τις δυνάμεις μας σε μάτια θέματα. Κύριε Πορκέζιο, Σε ό,τι αφορά το, το μπλοκάρισμα της εξόδου των μεταναστών. Μιλάμε για 65.000 πρόσφυγες και ποια είναι η προσέγγιση της Αυστρίας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας ε, τις τελευταίες εβδομάδες. το Σέγγεν, ε, ε, ο κανονισμός του Δουβλίνου προέρχονται από άλλες εποχές. Η δική μας προσέγγιση λοιπόν είναι οι αρχές να έχουν την επαφή με τους ανθρώπους και θα ήθελα να σας παραπέμψω στα λόγια του καγκελάριου Κούρτς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι την σημερινή μετανάστευση θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό μαζικής μετανάστευσης. Υπάρχει το θέμα της παγκόσμιας ασφάλειας, ε, του ε, χάσματος στα εισοδήματα. Ε, δεν είναι προβλήματα που εμφανίστηκαν ξαφνικά από το πουθενά. Εσείς από, ε, στην Ιταλία το ζήσατε αυτό από το 2011, εμείς στην Κεντρική Ευρώπη από το 2015. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε λοιπόν νέα εργαλεία, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εποχές παγκοσμιοποίησης. Η επόμενη ερώτηση ήταν του κυρίου Κάρας. Πού βρίσκεστε. ναι, τώρα σας βλέπω. Ναι. Δεν μιλώ μόνο για την Ιεμένη. Ε, όλοι οι πόλεμοι που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι ε, πόλεμοι ε, αντιπροσώπων ε, δεν είναι εμφύλιος πόλεμος, εκπροσωπούνται άλλα συμφέροντα εδώ. Και για την Γεμένη έχω ακούσει πολύ σοφά λόγια. Το Ιράν δεν ήταν πρόβλημα πριν τον Μάρτιο του 2015 που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Και η Γεμένη δεν βρίσκεται στο δικό μας ραμπάρ, ραντάρ. Συγγνώμη. Ε, πού πηγαίνουν οι πρόσφυγες, στη Σομαλία πάνε, δεν ε, περνάνε τη Μεσόγειο. Στο κέρας της Αφρικής πάνε για να επιβιώσουν. Η Γεμένη αποτελεί την πιο σημαντική ανθρωπιστική τραγωδία από το 1945, με όλο το σεβασμό για τα όσα έχουν συμβεί στη Συρία τα τελευταία χρόνια. Ναι, και στη Συρία βλέπουμε να εκτελήσεται ένα δράμα, στη Γεμένη όμως βλέπουμε καταστροφή. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών και με όσους προσπαθούν να, κάνουν, να πετύχουν κάποια πράγματα εκεί. Κύριε Κάρα, στο Κωσυφοπαίδιο. Ναι, την ώρα που θέτατε την ερώτηση σκεφτόμουν και εγώ ναι. Πόσο, πόσο δίκιο έχετε. Η μόνη απάντηση είναι να μιλάμε, να συζητάμε. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την διπλωματία και την εξωτερική πολιτική. Ε, ε, ε, με κανέναν τρόπο να μην διακόψουμε τις συνομιλίες. 21 Μαρτίου βρέθηκα στην ε, Πριστίνα, τα Σκόπια και το Βελιγράδι και ήταν ε, πολύ δυσάρεστο να παρακολουθούμε πόσο γρήγορα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα. Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει στις 12 η ώρα τι θα συνέβαινε στις 2.30 το απόγευμα. Θα πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε και να καλούμε τον κόσμο να επιδείξει πολιτική οριμότητα και ευαισθησία. Χρειάζεται ρεαλισμός. Πολυφωνία. Θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα και μου έχουν ξαναθέσει παρόμοιο ερώτημα και απάντησα ως εξής. Ο συντονισμός, η συνεννόηση είναι ένα θέμα. Για μένα πιο σημαντικό είναι όμως σε τι βαθμό όταν μιλάμε για, τις μεγάλες, για, για τα μεγάλα κράτη με μεγάλη ευθύνη, τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης, πώς προσεγγίζουν την εξωτερική πολιτική. Η προσωπική μου πείρα του τελευταίου εφτάμινου δείχνει ότι όλο και λιγότεροι υπουργοί πηγαίνουν στα συμβούλια. Έχουμε υψηλόβαθμους ε, αξιωματούχους, έχουμε πρέσβεις, αλλά είναι Συμβούλιο Υπουργών. Όλο και λιγότεροι λοιπόν βλέπουμε παρουσία των ε, υπουργών και οι αξιωματούχοι απλά αντιγράφουν τα παλαιότερα. Πολλούς ε, συναδέρφους μου δεν έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό είναι το θέμα. Πώς λοιπόν μπορώ να δείξω την ε, αφοσίωσή μου, την προσήλωσή μου στους στόχους σε πολιτικό επίπεδο. Κύριε Φρόιντ, εάν αποτελεί αρμοδιότητά μου η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ε, κυβερνητικό συνασπισμό της διαπραγματεύσεις του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου συνεχίστηκε αυτό που βλέπουμε σε πολλές πρωτεύουσες από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά. Συγκέντρωση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Καγκελάριου δηλαδή. Έτσι λοιπόν στην Αυστρία συνεχίσαμε μια παράδοση που γνωρίζουμε από άλλα Υπουργεία. Ε, δεν μου λείπουν τα θέματα αυτά, διότι έχω πάρα πολλή δουλειά στο γραφείο μου, ούτως ή άλλως. Ε, συμμετέχω στα Συμβούλια Εξωτερικών Υποθέσεων και πραγματοποιώ και πολλές διμερείς συναντήσεις. Ε, δεν έχω την εντύπωση ότι μου έκλεψε κανείς ε, κάποιο θέμα του χαρτοφυλακίου μου. Ε, έχω πράγματα να ασχοληθώ. Διατλαντική σχέση. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε σε ίσο επίπεδο. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια Ευρώπη με περισσότερη αυτοπεποίθηση, με περισσότερη συνείδηση. Κύριε Μέζεριτς, σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω, ουγγρικά δεν μπορώ να μιλήσω πολύ καλά. Όπως απάντησα και στην προηγούμενη μου ερώτηση, να συνοψίσω ως εξή. Τα μέσα που έχουμε, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών του Δουβλίνου, προέρχονται από τις εποχές πριν την παγκοσμιοποίηση υπολογίζαμε ε, ότι το πολύ 100 άνθρωποι θα ζητούσαν άσυλο. Σήμερα όμω έχουμε τελείως διαφορετική κατάσταση και γι' αυτό χρειαζόμαστε άλλα μέσα. Όσον αφορά τη Ρωσία. Η Ρωσία αποτελεί εταίρος σε πολλά θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πάνω στα θέματα αυτά έχοντας συνείδηση της γεωγραφίας. Και το τελευταίο θέμα, Ασία, Λατινική Αμερική. Δύο λόγια για την Λατινική Αμερική. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντήσω ξανά του συναδέλφου από τη Λατινική Αμερική. Κάποιου έχω ήδη ξανασυναντήσει στη Γενική Συνέλευση. Θα συμμεληθεί και το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Μιλάμε, θα πρέπει να μιλήσουμε, να θέσουμε ως προτεραιότητες, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Μιλάμε για μια μισή ήπειρο ε, εσείς έχετε άλλα συμφέροντα στη Λατινική Αμερική. Εγώ προέρχομαι από μια κεντροευρωπαϊκή χώρα, οπότε για μένα η Λατινική Αμερική είναι πιο πολύ νοτιοδυτική ε, σε σχέση με τη δική μου γεωγραφική θέση. Ε, λυπάμαι, αλλά ρεαλιστικά αυτό είναι η κατάσταση, η πραγματικότητα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στους επόμενους έξι μήνες θα εστιάσω πιο πολύ στα θέματα τα οποία σας ανέφερα. Αν θέλει κανείς να δει πραγματιστικά την κατάσταση, δεν μπορεί να είναι παρόν στη Λατινική Αμερική, την Κεντρική Αμερική, τόσο όσο και αλλού. Παρ' όλα αυτά, η υπηρεσία εξωτερική δράση λειτουργεί. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τη συνάντηση με τη ΣΕΛΑΚ, Γενική Συνέλευση. Εσείς αναφέρατε την Καράγου και τη Βενεζουέλα πιο συγκεκριμένα. Παρακολουθούμε την κατάσταση με πολύ προσοχή. Η Αυστρία δεν έχει πλέον πρεσβεία στο Καράκας, αλλά μέσω της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και αν τα γεγονότα το απαιτήσουν, θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαστε παρόντες. Όπως σας είπα θα αντικαθιστώ την Φεντερίκα Μογκερίνη όπου χρειάζεται. Δεν είδα να έχει κάποια παρουσία στην Λατινική Αμερική Φεντερίκα Μογκερίνη έτσι, με μια ματιά που έριξα. Αλλά αν χρειαστεί θα το κάνω και αυτό, θα είμαι παρούσα. Από προσωπικής πλευράς ε, η Λατινική Αμερική είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου. Αυτό έχω να σας πω. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή επιτυχία και ελπίζω ότι θα τα πούμε, ξαναπούμε σύντομα σε καλές συνθήκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ Κνάισελ, για αυτή τη συζήτηση. Πολύ καλή τύχη και καλή επιτυχία στην Αυστρία στο ρόλο του οικοδόμου ε, συνένεσης ε, σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών θεμάτων που μας απασχολούν. Θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συνάντησή μας. Ε, όσοι δεν ενδιαφέρεστε για τις εξελίξεις στο Μαυροβούνιο, παρακαλώ πολύ εγκαταλείψτε την αίθουσα για να συνεχίσουμε οι υπόλοιποι. Σε ένα λεπτό ξεκινάμε. So, ladies and gentlemen, we're 20 minutes. Ήδη έχουμε μια καθυστέρηση 20 λεπτών. Περνάμε στο σημείο 5 σημεία τη διάταση. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο. Μετά τη Σερβία, το Κοσμοπέδιο και την Αλβανία που συζητήσαμε τον Ιούνιο, τώρα περνάμε σε αυτή τη χώρα, το Μαυροβούνιο. Το έχει οριστεί από τον πρόεδρο της Κομισιόν ως ενδεικτική ημερομηνία μέχρι την οποία το Μαυροβούνιο και ενδεχομένως και η Σερβία θα μπορούσαν να έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ως κίνητρο περισσότερο προκειμένου να συνεχίσουν το δρόμο των μεταρρυθμίσεων που θα τους οδηγήσει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει 31 από τα 35 κεφάλαια, πρωτοπορεί. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζει σημαντικέ προκλήσεις σε θέματα όπως η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η διατήρηση ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Δίνω το λόγο στον κύριο Τσάλ Στάνο, τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαδικασία του Βερολίνου και το φορμάτ ε, λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο σχεδόν ταυτόχρονα. Πάμε βέβαια που ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μου δεν κατάφερε να παραστεί χτες. Δείχνει ενδεχομένω όμως αυτή η συνεδρίαση ότι το Ηνωμένο θέλει να παραμείνει στα Δυτικά Βαλκάνια ισχυρό παίκτη. Είμαι εισηγητή για το Μαυροβούνιο εδώ και 8 χρόνια. Έχω προσπαθήσει να βρω την ορθή ισορροπία ανάμεσα στου επένου για την πρόοδο και τι ε, παρατηρήσει σε ό,τι αφορά τα σημεία στα οποία χρειάζεται βελτίωση. Το Μαυροβούνιο είναι η χώρα που έχει προχωρήσει περισσότερο. 31 ε, ανοιχτά κεφάλαια από τα συνολικά 35 του κοινοτικού και Περιμένουμε πιο πολλά πράγματα από το Μαυροβούνιο λοιπόν από ό,τι από τους υπόλοιπους. Και έχουμε βάλει πιο ψηλά τον πύχια. Από την προηγούμενη έκθεσή μας Λαμαχώρα χώρα προεδρικές εκλογές, συγχαρητήρια στον πρόεδρο Βουκάνοβιτ. Η έκθεση του ΟΑΣΕ ανέφερε ότι οι εκλογές σε σύμφωνα με τα δημοκρατικά πρότυπα. Έχουν επανέλθει σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα στο Κοινοβούλιο πλέον, μετά από ένα μποϊκοτάζ, μερικό μποϊκοτάζ που είχε ξεκινήσει από το 2016. Είναι σημαντικό και τα υπόλοιπα κόμματα να επιστρέψουν ανεφόρων στο Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου. Οι συστάσεις του ΟΑΣΕ για τις ε, μελλοντικές εκλογές θα πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν οι πολιτικοί έχουν τη θέση τους στο Κοινοβούλιο και τη χρησιμοποιούν. Στην έκθεση εστιάζουμε στην ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του τύπου και των μέσων ενημέρων. Ε, το θέμα με το RTCG, το Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Οργανισμό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Για, είναι μια ευκαιρία να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές και μια ευκαιρία για την κυβέρνηση να δείξει ότι είναι προσιλωμένη στην ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Είναι μια χρονιά που είδαμε ε, την Ολιβέρα Λάκιτς να ε, δέχεται επίθεση με πυροβολισμό στο πόδι και, μια, και ένα άλλο δημοσιογράφο, τον κύριο Σαντίκοβιτς, να βλέπει το, ένα παγιδεμένο αυτοκίνητο να κρίνεται μπροστά στο σπίτι του. Επιθέσει λοιπόν εναντίον της ελευθερίας του τύπου. Ε, ήταν και οι δύο δημοσιογράφοι που ασχολόντουσαν με υποθέσεις οργανωμένου κλίματος και διαφθοράς. Αυτές οι περιπτώσεις είναι προφανώς ακραίες. Αναγνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του έτους μόνο εννέα τέτοιου είδου επιθέσει ή εκφοβισμοί έλαβαν χώρα. Αλλά και πάλι και εννιά πολλοί είναι εναντίον δημοσιογράφων. Πολλέ είναι εναντίον δημοσιογράφων. Αυτά συνδέονται με την έκκλησή μα να αναλυφθεί περισσότερη δράση κατά τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο. Ήδη το Μευροβούνιο έχει δείξει καλή διαγωγή σε αυτό το θέμα και ελπίζουμε θα συνεχίσει. Ελπίζω θα ξανα θα δούμε ε, να εφαρμόζεται το καινούριο σύστημα διορισμού των ανώτερων δικαστικών. Τέλος, δύο λόγια για την ε, δίκη του, ε, της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016. Δεν θα σχολιάσω οποιαδήποτε λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά την τρέχουσα ακροματική διαδικασία, αλλά η διαδικασία αυτή είναι ορθή, Όλες οι ακροάσεις είναι δημόσιες. Τέτοιου είδου δικαστική διαφάνεια θα αποτελέσει πρότυπο για το μέλλον. Πολύ σημαντικό αυτό προκειμένου να αντιμετωπιστούν δια, ε, θεωρίες συνωμοσία. Το Μαυροβούνιο θα πρέπει να παραμείνει στο σωστό δρόμο, σωστή άγουσα. Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδό του και νομίζω ότι μόνο ο χρόνος είναι ότι ο χρόνος είναι το μόνο εμπόδιο στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου. Θα περιμένω τα σχόλιά σας και ελπίζω ότι θα μπορέσω να διευκρινίσω οποιαδήποτε θέματα είναι αόριστα ή οποιαδήποτε παραλήψεις έχουν γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Τώρα θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο στον David Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν δεν σας πειράζει, ο κύριος Άντριο Λάκη κύριος Ανδρουλάκης θα ήθελα, ε, δεν είναι εδώ, θα ήθελα να μιλήσω εξ Πρώτα απ' όλο ο κύριος Ανδρουλάκης θα ήθελε να ευχαριστήσει τι ευχαριστίες του στον κύριο Τάνακ για όλη τη δουλειά του και τη συνεργασία του. Είναι πραγματικός φίλος του Μαυροβουνίου και θα μας λείψει. Κατά τη διάρκεια της παρουσίαση της στρατηγική της Κομισιόν για την συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια, ε, ε, διαπιστώσαμε ότι δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει χρόνος για να κλείσουμε παραπάνω κεφάλαια διαπραγμάτευσης. Και μέχρι το 2025 το Μαυροβούνιο μπορεί να γίνει το 28ο κράτος μέλος. Ο κύριος Ανδρουλάκης συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσης σχετικά με τις βελτιώσεις που είναι απαραίτητες στο τομέα του κράτους δικαίου μεταξύ άλλων και ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις και να ε, προαχθεί η κοινωνική ασφάλεια. Επίσης, η καταπολέμηση των ε, διακρίσεων ε, στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να πω και λίγα λόγια ως ε, Πρόεδρος της Επιτροπής Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πλήρη έκθεση. Τα περισσότερα στοιχεία θα μας χρησιμεύσουν ε, για τα, ε, τις που θα παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ καλά νέα αυτά που μας λέτε και κυρίως το θέμα της επιστροφής ενός μέρους της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ε, κόμματα που είναι υπέρ της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές, θα είμαι πιο... Ε, θα ασκήσω μεγαλύτερη κριτική. Υπάρχει θέμα με τις θεμελιώδεις ελευθερίες. δεν έγιναν ε, τηλεοπτικές αναμεταδόσεις ε, συζητήσεων και δεν ε, είχαν την ευκαιρία οι ψηφοφόροι να κάνουν επιλογές με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και δηλώσεις. Αυτά αναφέρει μία έκθεση. Χρειάζονται λοιπόν μεταρρυθμίσεις στο τομέα των εκλογών Ελπίζω με την επιστροφή της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να κάνουν μία πρόοδο σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου και τις σχετικές ανησυχίες. Θα ήθελα να πω, πρόκειται για τομέα ότι δεν έχει γίνει καμία πρόοδος σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες σε αυτό το τομέα. Υπάρχει κάτι που δεν αναφέρθηκε στην έκθεση και αξίζει να σημειωθεί. Ε, οι τιμές των ακινήτων. Οι αρχές στο Μαυροβούνιο ε, κάνουν αυθαίρετη χρήση πολιτικής ε, απαλωτρίωσης και δεν υπάρχει έννοια της ε, προσωπικής ιδιοκτησίας στο Σύνταγμα του Μαυροβουνίου. Υπάρχει μια πολύ αόριστη αναφορά Πρέπει λοιπόν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Ε, κάποιοι έχασαν τις ιδιοκτησίες τους ε, υπό το κομμουνιστικό καθεστώς του παρελθόντος, αλλά η πρόοδος είναι πολύ αργή. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το Μαυροβούνιο κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και πολύ σωστά σημειώσατε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και ε, η έκθεσή σας ήταν ιδιαίτερα πλήρης. Ευχαριστώ. Martin, for your... Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρτιν. Εξ ονόματος του ε, S&D και της αντιπροσωπεία Αντιπροσωπείας Σταθεροποίησης και Συμφωνίας Σύνδεσης, το ε, ΕΛΚ εκπροσωπείται από τον κύριο Πέτερλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλο τον κύριο Τάνοκ για την εξαιρετική έκθεση που βασίζεται σε ρεαλιστικά και πραγματικά στοιχεία για την κατάσταση στο Μαυροβούνιο. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Δεν θα επαναλάβω όσα έχουν πει προλελήσεντες σε ό,τι αφορά τους τομείς στους οποίους είναι απαράτητη περαιτέρω πρόοδος. Για μία ακόμη φορά υπάρχει περιθώριο πρόοδου και γι' αυτό το λόγο η αξιολόγηση ε, ε, ήταν καλύτερη στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης. Ε, προχώρησαν σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των συνόρων με το Κωσυφοπαίδιο και γι' αυτό το λόγο με εκπλήσει το γεγονός ότι διαβάζουμε στην έκθεση ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα των συνόρων με άλλες χώρες. Η... Αναφέρθηκε σε αυτό και η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας. Ε, η αντιπροσωπεία μας θα είναι επί τόπου την ερχόμενη εβδομάδα και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτερλε. Εξ ονόματος της ομάδας Άλντα, ο κύριος Ράντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τάνοπ για αυτή την εξαιρετικά ισορπημένη έκθεση. Τα τελευταία χρόνια το Μαυροβούνιο σημείωσε σημαντική πρόοδο. όμως σε κάποιους σημαντικότατους τομεί δεν έχει σημειωθεί καθόλου πρόοδο. κυρίως σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερου τομεί. και αυτό δείχνει, η ελευθερία τύπου δείχνει την ε, δημοκρατική ισχύ ενό ε, κράτους σε διάστημα κάποιων ετών δεν σημειώθηκε ε, καμία πρόοδος. Ασκήθηκαν πιέσεις ε, εις βάρος ε, δημοσιογράφων, περιπτώσεις εκφοβισμού τα τελευταία χρόνια. Το Μαυροβούνιο υιοθέτησε σημαντικούς νόμους σχετικά με τη χρηματοδότηση ΜΚΟ, της, ε, των τηλεοπτικών καναλιών, όλα αυτά καθιστούν μια ε, πολύ σημαντική δημοκρατική υποδομή. Όμως, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την εφαρμογή αυτών των των νόμων, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι είναι εύκολη η θέωτηση ε, νόμων, αλλά με την εφαρμογή τι γίνεται και με τις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις ε, υπάρχει πρόβλημα με τη διαφθορά. Εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την, το άνοιγμα του κεφαλαίου 25 σχετικά με το κτηματολόγιο, την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο ε, στον τομέα των επιχειρήσεων στο Μαυροβούνιο και για να έχει πρόσβαση το κοινό ε, στην ε, πληροφόρηση και στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών είναι σημαντικότατες οι ψηφιακές τεχνολογίες. Για μία ακόμη φορά, ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνο για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Η πράσινη, ο κύριος Μέζεριτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ για το σχέδιο έκθεσής του. Είναι πράγματι πολύ καλό και ισορροπημένο κείμενο. Ίσως επειδή είναι μια από τις πιο εύκολες υποθέσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως και να έχει όμως, είναι τέχνη το να εκπονήσει κανείς μια ισορροπημένη έκθεση. Συγχαρητήρια λοιπόν. Τούτου λεχθέντος δεν θέλω να μακρηγορήσω μιλώντας για την πρόοδο που βλέπουμε και ενθαρρύνουμε στο Μαυροβούνιο. Είμαστε ικανοποιημένοι με την ε, γενική ανάπτυξη και τον προσανατολισμό ε, προς το στόχο της προσχώρησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουμε το να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, θα ήθελα να φέρω κάποια θέματα. Στην παράγραφο 7, ο εισηγητής πολύ σωστά λέει ότι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία είναι η ε, υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Υπάρχει ένας ε, πολύ επαγγελματία διευθυντή ΜΚΟ, μέλος του Συμβουλίου, που απολύθηκε και δεν είναι η μόνη περίπτωση μη κυβερνητική οργάνωσης ε, που παραμερίζεται στο περιθώριο. Δεν λέμε ότι είναι γενική τάση, αλλά είναι ανησυχητικό περιστατικό και θα θέλαμε πολύ να επανεξεταστεί στο βαθμό που είναι δυνατό από την κυβέρνηση. Επίσης, καταπολέμηση της διαφθοράς με αποτελεσματικό τρόπο και μιλώ εκ πείρας. Απαιτείται διαφάνεια σχετικά με το πώς δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια. Δεν ε, τα πάνε πολύ καλά και όλα τα κράτη-μέλη στο θέμα αυτό. Λυπούμαστε όμως που με τις νέες νομοθετικές αλλαγές του Ιουνίου βλέπουμε μείωση της διαφάνειας σε πολλά θέματα όπως είναι για παράδειγμα οι πληροφορίες ε, για την ε, δημιουργία δρόμων ε, και πληρωμές από τον προϋπολογισμό κατά την προεκλογική περίοδο. Και αυτή η τάση θα πρέπει να αντιστραφεί εάν η κυβέρνηση θέλει στα σοβαρά να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Θα πρέπει η διαφάνεια λοιπόν να αποτελέσει προτεραιότητα. Όσον αφορά το περιβάλλον, στηρίζουμε την θετική διατύπωση στην παράγραφο 29 για την τοποθεσία Ούλζιν Σαλίνα και πιστεύουμε ότι θα χρειαστούν μελέτες αντικτύπου. Κάθε φορά που υποβάλλεται σχετική έκθεση εμείς υποβάλλουμε τροπολογίες. Και το πρόγραμμα στον ποταμό Μωράτσια επίσης ε, θα πρέπει να επανεξεταστεί όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επίσης, όσον αφορά την ομάδα ε, παρακολούθησης των εκλογών, Συμφωνώ με την έκθεση του ΟΑΣΕ, αλλά θα ήθελα να πω ότι το θέμα δεν είναι αυτό που, γίνεται την ημέρα των εκλογών όσον αφορά το πόσο δίκαιες και διαφανείς είναι οι εκλογές. Όλη η προεκλογική περίοδος μας ενδιαφέρει. Και όχι μόνο η προεκλογική περίοδος. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε αποτελεσματικά εργαλεία για αξιολόγηση και αυτής της περίοδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Χατζηγεωργίου από τους Πράσινους. Thank you, Mr. President. I don't have many things... Δεν έχω και πολλά να πω. Το Μαυροβούνιο έχει προχωρήσει πολύ στην διαδικασία προσχώρησης. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τάνοκ για την ισορροπημένη του έκθεση. Είναι πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Το Μαυροβούνι βέβαια έχει ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει προκειμένου να γίνει πλήρες μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο ότι συμφωνώ με τον κύριο Μέστεριξ ότι και άλλε χώρε αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Τη διαφθορά, για παράδειγμα, η διαφθορά είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για μας ο σεβασμός στα κριτήρια της Κοπεχάγης, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σημαντικό πρόβλημα για αυτή τη χώρα. Ο τρόπος που δαπανώνται τα κρατικά κονδύλια, που θα πρέπει να είναι όσο πιο αποτελεσματικός γίνεται. Και τέλος, να πω όλα αυτά ότι στην έκθεση Φίσταται και μία φράση για την είσοδο του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ. Κατά την άποψή μας, μια χώρα η οποία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοδοξία της ίδιας χώρας ενδεχομένως να εισέλθει να ενταχθεί σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Η FTD δεν είναι παρούσα, ούτε η NF, ε, μία εγγεγραμμένη, όχι κανένας. Ένας ακόμη ε, ομιλητής έχω, είναι στον κατάλογο μου και ο Σπίτσουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση Τάνοκ είναι πολύ ισόρροπο έγγραφο εντοπίζει τα σημεία στα οποία το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει πρόοδο και ταυτόχρονα εντοπίζει τα πιο σοβαρά προβλήματα της χώρας. Για παράδειγμα, αυξημένος αριθμός πολιτικών δολοφονιών, δράση του οργανωμένου εγκλήματος που επηρεάζει την ασφάλεια των πολιτών κλπ. Απειλές εναντίον του τύπου, επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων. Από την άλλη μεριά, έχει σημειωθεί συνολική πρόοδος. Έχουν ανοίξει 31 από τα 35 κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου. Κάτι που καθιστά το Μαυροβούνιο επικεφαλής της ομάδας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές χαρακτηρίστηκαν από ελάχιστε παρατυπίες, θα πρέπει να διορθωθούν. Το Μαυροβούνιο στηρίζει την περιφερειακή συνεργασία και σύντομα θα πρέπει να λύσει και τα συνοριακά του προβλήματα με τους γείτονες. Η Ποντγκόριτσα στηρίζεται και από το Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν, αλλά πριν το Μαυροβούνιο ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα αριθμό θεμάτων που έχουν σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για αυτό το λόγο η κυβέρνηση θα πρέπει να διατηρήσει το διάλογο με την κοινωνία και η συνολική πρόοδος σίγουρα θα επηρεαστεί από τις σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση επιστρέφει σιγά σιγά και αυτό πρέπει να το κολοσορίσουμε. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτσουλα. Άλλοι συνάδελφοι θα ήθελαν το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης. Νιερ. Δεν σας βλέπω. Κυρία Κρυμμένο. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τάνοκ, αγαπητά μέλη, να σχολιάσω ε, συγγνώμη, να επενέσω καταρχήν τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τη γενική σας ε, κρίση σε ό,τι αφορά την πρόοδο του Μαυροβουνίου. Η έκθεσή σας αναφέρεται στην προσήλωση της Κομισιόν σε όλη την περιοχή. Σύμφωνα με την ε, δήλωση για τα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες τις οποίες και υλοποιούμε. Το Μαυροβούνιο είναι η χώρα που πιο πολύ έχει προχωρήσει, 31 κεφάλαια ανοιχτά, 3 έχουν κλείσει προσωρινά. Το τελευταίο που άνοιξε είναι το κεφάλαιο 17, οικονομική και νομισματική πολιτική και άνοιξε στις 25 Ιουνίου. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με βάση την πρόοδο που θα έχει πετύχει το Μαυροβούνιο. Όμως, περαιτέρω πρόοδο θα επιτευχθεί μόνο αν το Μαυροβούνιο δώσει προτεραιότητας, το κράτος δικαίου, μεταξύ, ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, του ξεπλήματος ε, χρήματος, χρημάτων και, και επίσης στον αγώνα για να αντιμετωπιστούν να αντιμετωπιστεί η βία εναντίον δημοσιογράφων και τα προβλήματα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κεφάλαια 23 και 24, τα κεφάλαια 23 και 24 θα εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζουν, να χαρακτηρίζουν τη συνολική πρόοδο του Μαυροβουνίου. Τέλος, ενθαρρύνουμε όλους τους πολιτικούς φορείς στο Μαυροβούνιο να αποκλιμακώσουν τη συνένταση και να ξαναφέρουν το διάλογο στο Κοινοβούλιο. Με την σταδιακή επιστροφή των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο βλέπουμε να γίνεται ένα πρώτο βήμα το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Είμαι πεπισμένη ότι τα συνεχή και συνεπή μηνύματα που προέρχονται και από το Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν θα δώσουν στο Κοινοβούλιο επαρκή όθηση προκειμένου να παραμείνει αξιόπιστο στο δρόμο προς την ένταξη. Ευχαριστώ πολύ μια ακόμα φορά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το ψήφισμα και για την αξιόλογη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι. Δίνω και πάλι το λόγο λοιπόν στον κύριο Τάνο. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πολύ για τα θερμά λόγια και την ενθάρρυνση που άκουσα από τους συναδέλφους από όλο το πολιτικό φάσμα στην Επιτροπή μας. Πράγματι, μέχρι το 2025 το Μαυροβούνιο θα είναι να γίνει μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με εκπλήσει το γεγονό ότι ως σοσιαλιστής αναφέρθηκε ε, στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Αναφέρθηκε ε, και στη διεξαγωγή των εκλογών, στις, στην ανεπάρκεια πολιτικής συζήτησης και στην επαρκή, στον επαρκή αριθμό υποψηφίων. Επίσης, το θέμα της οριοθέτησης των συνόρων με την Κροατία. Έχω αναφερθεί σε αυτό το θέμα σε προηγούμενη έκθεση. Η ελευθερία του τύπου ε, αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα δεν μίλησα συγκεκριμένα για το εκτιματολόγιο και το κεφάλαιο 25. Φυσικά θα καλωσορίσω ε, οποιαδήποτε πρόοδο σε αυτό το τομέα. Ο κύριος Μέζερης εξ των Πράσινων ε, αναφέρθηκε στην καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Θα χρειαστώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση της διαφάνειας ε, και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Στο παρελθόν με την κυρία Λούνατσεκ συζητήσαμε επί μακρόν για το κατά πόσο ε, αναφέρεται το θέμα του περιβάλλοντος στις εκθέσεις μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζιογεωργίου σε ό,τι αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ. Πράγματι ε, παλιά ε, διαμάχη με πολλά ε, μέλη τα τελευταία χρόνια. Δέχομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι δύο διαφορετικά θέματα. Όμως πρόκειται για πολυμερείς οργανισμούς που προσπίζονται τις κοινέ αξίες μας και τη δημοκρατία μας. Και αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει απειλέσεις. Άρα πρέπει να ε, χαιρετήσουμε το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο ε, θέλει να κατευθυνθεί σε αυτό, προς αυτό το... Ε, πρέ, θέλει να λάβει αυτή την κατεύθυνση και είναι μέλος του ΝΑΤΟ πλέον. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. 31 Αυγούστου, 11 η ώρα η προθεσμία για την απολογή τροπολογιών. Η ε, ε, ψηφοφορία θα γίνει 8 ε, ή 9 Οκτωβρίου στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτο 2019, όλα τα τμήματα. Να υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνια, κάθε ε, φορά, κάθε έτος μιλάμε για δύο διαφορετικά θέματα. Πρώτα όλα θα υποβάλουμε τροποποίηση στο σχέδιο προπολογισμού που παρουσίασε η Κομισιόν και δεύτερον θα υιοθετήσουμε μια γνωμοδότηση σχετικά με το ε, ψήφισμα που θα ε, συνοδεύει το προπολογισμό. Θα ακούσουμε τον εισηγητή σχετικά με τις πιθανές ε, τροπολογίες μεταξύ άλλων. Αγαπητέ συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Προπολογισμών μου που συνεργάστηκε με την Επιτροπή ΑΦΑΤ και έλαβε υπόψη πολλές από τις ανησυχίε μας σε αυτή την ε, έκθεση. Βρισκόμαστε σε ένα ε, σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά τη συμβολή μας ε, στο προϋπολογισμό. Σήμερα συζητάμε το θέμα της γνωμοδότησης. Ε, ε, προβλέπουμε ήδη την τοποθέτηση του Συμβουλίου που θα αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά το κείμενο της ε, Κομισιόν, βλέπουμε τις παλιές κακές συνήθειες που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια. Ε, περικοπές, για να ξενοικονομηθούν. κονδύλια. Εμεί θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, για να επιμείνουμε ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την εξωτερική της δράση. Χρειάστηκε να εστιάσουμε το κείμενο στις σημαντικότερες προτεραιότητες. Ανησυχήσαμε για το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στον τομέα 4 ε, αντιπροσώπευε κυρίως τη διάθεση κονδυλίων για την εφαρμογή της συμφωνίας με τη Τουρκία. Χρειάζονται επίσης περισσότερα κονδύλια για τα Δυτικά Βαλκάνια, δεδομένης της στρατηγικής που δρομολογήθηκε το περασμένο Φεβρουάριο. υπάρχει και το, ο μηχανισμός προνταξιακής βοήθειας 2 ε, και η ανάγκη να ε, να δοθούν κονδύλια στην ε, κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση του δεύτερου ε, τμήματος του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στα πλαίσια της συμφωνίας με τη Τουρκία ε, ένα δισεκατομμύριο η, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν δύο δισεκατομμύρια τα κράτη-μέλη. Επίσης αναφέραμε το γεγονός ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη βοήθεια που δίνουμε στην ε, την Ισία και τη Λιβύη. Πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως ό,τι αφορά τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν όλα ένα και μεγαλύτερες πιέσεις και πρέπει να ε, ανανεώσουμε την υποστήριξή μας στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και φυσικά τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσω διάφορες τροπολογίες προκειμένου να συμπληρωθεί αυτό το ε, κείμενο και θα ε, λάβω υπόψη κάποια σημεία που αναφέρονται στο γράμμα που στείλετε στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και θα χαρώ να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πενιφέη. Φτάνουμε στους ομιλητές που έχουμε στο κατάλογό μας. Μόνο ένας συνάδελφος έχει ζητήσει το λόγο. Δύο. Δίνω καταρχάς λοιπόν το λόγο στον μοναδικό Νταν Christian Πρέντα. Euh, Διαπιστώβω ότι πέντε μέλη είναι παρόντα, συνολικά. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές. και φέρα την έκθεση Μπενιφέη. θέλω να τον συγχαρώ καταρχήν. Συμφωνώ εν γέννη με τον τρόπο που διαβάζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το τμήμα 4. Η αύξηση είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Παρ' αυτά, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η αύξηση ε, αφορά περισσότερο την στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία. Και μάλιστα θα μας μείνει πολύ λίγο περιθώριο ελιγμού του χρόνου σε περίπτωση κρίσης ε, είτε στη γειτονιά μας είτε αλλού στον κόσμο. Με ανησυχεί ιδιαίτερα η μείωση των ποσών για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι στην προσήλωσή μας στην περιοχή αν μειώνουμε τη χρηματοδότηση. Με περικοπές δηλαδή του προπολογισμού που αφορά αυτή την περιοχή. Είναι σημείο κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης. Επιπλέον, με ανησυχή, η πιέση που δέχεται το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας. Θα ήθελα να αυξηθεί επίσης το Ταμείο κοινή Πολιτικής Ασφάλειας που είχε μειωθεί στο προσχέδιο της Κομισιόν. Θα πρέπει επίση να στηρίξουμε όλα τα μέσα που έχουν σχέση με τη σταθερότητα και την ειρήνη και να υπογραμμίσουμε την σημασία να έχουν επαρκείς πόρους. Θέλω να χαιρετήσω την ένταξη του προγράμματος για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα που θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στο, στα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά την εδραίωση μιας ευρωπαϊκής άμυνας. Ε, είμαι πεπισμένος ότι ως και ως ηγητής στους επόμενους μήνες θα συνεργαστώ με τον κύριο Μπονιφέη και ότι όλα όσα μόλις σας ανέφερα τελικά θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο της έκθεσης. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Σαπίνε Λούιζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι θα μιλήσω γερμανικά και θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους γερμινείς, λέει η ομιλήτρια, που σήμερα βρίσκονται στην 36η μέρα της διαμαρτυρίας τους. Κύριε Μπενιφέη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε με την γνωμοδότησή σας ιδιαίτερα όσον αφορά την διευκόλυνση με την Τουρκία. Συμφωνούμε με αυτά που γράφεται στη γνωμοδότηση. Ωστόσο, βλέπουμε γενικά επικριτικά τα, τα πιστευματικά ταμεία και λόγω διαφάνειας, αλλά και όσον αφορά το τι θα χρηματοδοτηθεί από αυτά. Ιδιαίτερα όσον αφορά το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική. Το σημείο 7 της νομοδότησής σας με βρίσκει σύμφωνη. Λέει ότι πρέπει να ε, στηρίξουμε περισσότερο τις ζώνες σύγκρουσης. Αλλά η ερώτησή μου είναι μόνο κονδύλια λείπουν ή μήπως λείπει και η σωστή κατεύθυνση στην πολιτική. Για παράδειγμα, η Ουκρανία δεν θα ορθοποδήσει με νεοφιλελεύθερες πολιτικές, πόσο μάλλον αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά η διαφθορά. Η Τινησία, την οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την έχει ε, δαπανίσει προς όφελος της χώρας. Και στην Λιβύη χρειάζεται διαμεσολάβηση. Δεν χρειαζόμαστε εξαγωγές όπλων. Είναι ντροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία να μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα ενώ στην Βόρεια Αφρική να κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε μακριά τους ανθρώπους αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λουίζινγκ. Συνάδελφοι, υπάρχει άλλος που θα ήθελα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι ο κύριος Πενιφέη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι μια σαφής έκθεση και αποτελεί πολύ καλή βάση. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Είναι εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο συνάδελφος Πενιφέη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Δίνω το λόγο στον κύριο Μάρκ Τζόνσον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΕΡ. Πού βρίσκεστε, καλώς ήρθατε. Βρετανός ή Ιρλανδός είστε, Ιρλανδός είμαι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Η παρουσίαση αυτής της νομοδότησης ε, πραγματοποιείται σε πολύ ε, χρήσιμη στιγμή όσον αφορά τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο προχωράει στην εξέταση του προϋπολογισμού και αύριο στην Κορεπέρ θα γίνει συζήτηση και διαμόρφωση θέσης για το σχέδιο προϋπολογισμού που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο θέματα προκύπτουν από τη συζήτηση στο Συμβούλιο και που θα συμπεριληφθούν και στη, στο επόμενο στάδιο της συζήτησης του σχεδίου προϋπολογισμού εδώ ε, τα Δυτικά Βαλκάνια που αναφέρθηκαν αρκετέ φορές και φυσικά και η Τουρκία. Όσον αφορά την Τουρκία, θα ήθελα, επειδή είναι κάπως δύσκολο να αποκωδικοποιήσει κανείς ε, τα έγγραφα αυτά, θα ήθελα να διασαφηνίσω την πρόταση που έχουμε υποβάλει και να σας ενημερώσω σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις εντός του Συμβουλίου. Όσον αφορά την ε, κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού όπου θα προβλεπόταν ένα σημαντικό ποσό προς την Τουρκία φέτος. Πέρσι είδαμε εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν σε μείωση κατά 75 εκατομμύρια του ποσού που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προϋπολογισμό του 2018. Το σχέδιο προϋπολογισμού λοιπόν πέρσι τελικά οδήγησε σε 175 εκατομμύρια λιγότερα για την Τουρκία από ό,τι είχαμε προτείνει. 105 εξ αυτών χρησιμοποιήθηκαν οι άλλους ε, στόχους, ενώ το 70% ε, μπήκε στο αποθεματικό. Ενώ 70 ε, εκατομμύρια μπήκαν στο αποθεματικό. Και σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΠΑ, οδηγηθήκαμε σε επιπλέον μείωση των πόρων προς τη Τουρκία, σε 78 εκατομμύρια λιγότερα. Το οποίο σημαίνει ότι συνολική μείωση για την Τουρκία για το 2018 ανέρχεται σε 253 εκατομμύρια. Προσέξαμε λοιπόν τη θέση του Κοινοβουλίου την περσινή για τον προϋπολογισμό του 2018. Ο Επίτροπος Χάν βρέθηκε εδώ για τον στρατηγικό διάλογο για αναθεώρηση των εγγράφων της στρατηγικής και αναφέρθηκε ότι θα γίνουν περαιτέρω μειώσει. Και ουσιαστικά αυτό κάναμε όσον αφορά την Τουρκία στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Εάν λοιπόν είχαμε δει πού βρισκόμαστε όσον αφορά τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, κανονικά θα προτείναμε για την Τουρκία 650 εκατομμύρια ευρώ, κάτι λιγότερο από 650 εκατομμύρια. Ενώ τελικά για την Τουρκία προτείνουμε, εάν αφαιρέσουμε το ποσό για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες, που είναι σημαντικό θέμα, το ποσό είναι 252 εκατομμύρια λιγότερα, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε καθαρό ποσό σε όλες τις γραμμές του υπροπολογισμού για την Τουρκία, κάτι λιγότερο από 400 εκατομμύρια. Αναφέρθηκα στις γραμμές του προϋπολογισμού και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ανοίξω εδώ μια μικρή παρένθεση. διότι οι πόροι που έχουμε για την Τουρκία κατανέμονται σε τρεις βασικές γραμμές του προϋπολογισμού. Δύο γραμμές του υπροπολογισμού εμπίπτουν στον τίτλο 22, την ε, πολιτική γειτονίας. Ε, στήριξη για πολιτική μεταρρύθμιση και ευθυγράμμιση με το, κεκτημένο, το κοινοτικό κεκτημένο. Η δεύτερη είναι στήριξη για εδαφική ανάπτυξη και μετά έχουμε μία τρίτη γραμμή του προϋπολογισμού ε, στο τμήμα που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη, υποστήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη. Μιλάμε δηλαδή για ανάπτυξη της υπαίθρου για τις ε, χώρες προσχώρησης. Πέρα λοιπόν από τη μείωση κατά 253 εκατομμύρια στην πρότασή μας σε σχέση με το δημοσιονομικό προγραμματισμό και το, στρατη... και το έγγραφο ενδεικτικής στρατηγικής, σε επίπεδο ομάδας εργασίας υιοθετήθηκε θέση που ε, πιστεύω ότι θα υιοθετηθεί και από το Συμβούλιο. Η πρόταση λοιπόν της ομάδας εργασίας προβλέπει περαιτέρω μείωση για την Τουρκία κατά σχεδόν 147 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση αυτή συγκεντρώνεται αποκλειστικά στην πρώτη γραμμή του προϋπολογισμού που ανέφερα, δηλαδή υποστήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κεκτημένο, με το ενωσιακό κεκτημένο. Εάν αυτή τελικά είναι η οριστική θέση στον προϋπολογισμό, θα έχουμε κάποια προβλήματα, διότι αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού είναι η γραμμή μέσω της οποίας στηρίζουμε την συμμετοχή της Τουρκίας σε ενωσιακά προγράμματα όπως είναι το Εράσμους, το Φισκάλις, τα Τελωνία, την καταπολέμηση των ναρκωτικών, την επιβολή του νόμου και την υποστήριξή μας προς την κοινωνία των πολιτών. Το εισιτήριο λοιπόν για αυτά τα κοινοτικά προγράμματα πληρώνεται από αυτά τα κονδύλια. Και η υποχρέωση καταβολής αυτού του εισιτηρίου είναι διεθνής. Θεσπίζεται σε διεθνείς συμφωνίες ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν συμφωνίες που πρέπει να τηρήσουμε. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ανησυχητική η πρόταση του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εάν το Κοινοβούλιο δεν αντιστρέψει την πρόταση αυτή σε επίπεδο Συμβουλίου, εάν δεν αποκατασταθεί το σχέδιο προϋπολογισμού, θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση και κατά τη συνδιαλλαγή δεν θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Εάν από την άλλη, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν πολλές απόψεις για το θέμα αυτό, το Κοινοβούλιο θέλει να μειώσει τον προϋπολογισμό προς την Τουρκία για το 2019, θα ήθελα να σας επισημάνω τις γραμμές στις οποίες θα πρέπει να γίνει αυτό, διότι η μείωση αυτή τη στιγμή γίνεται στη γραμμή ακριβώς που πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση στην Τουρκία. Το άλλο θέμα που ήθελα να φέρω έχει να κάνει με τα Δυτικά Βαλκάνια. Όταν μειώσαμε ε, της, ε, την βοήθεια προς την Τουρκία κατά 253 εκατομμύρια, πήραμε τα χρήματα αυτά και τα βάλαμε στα Δυτικά Βαλκάνια. Εάν λοιπόν συγκρίνουμε τα στρατηγικά έγγραφα και τον ε, δημοσιονομικό προγραμματισμό που είχαμε πριν ένα χρόνο με αυτό που προτείνεται για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019, υπάρχει καθαρή αύξηση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή τα κονδύλια αυτά έχουν τοποθετηθεί στα προγράμματα πολλών κρατών. Στον δημοσιονομικό προγραμματισμό είχαμε 189 εκατομμύρια ευρώ για πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Στην περσινή διαδικασία του προϋπολογισμού ε, αυξήθηκε το ποσό αυτό κατά 10 εκατομμύρια ευρώ για φέτος. Και ουσιαστικά η μείωση Όπω γίνεται αντιληπτή, είναι μείωση σε σχέση με την αύξηση που είχε γίνει πέρσι. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο βασικές μου παρατηρήσεις. Θα ήθελα στην Επιτροπή σας να πω ότι φυσικά η Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ είναι διατεθειμένη να σας παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη, εξηγήσει για την πρότασή μας που μπορεί να επιθυμούν οι βοηθοί σας. Πολύ ευχαριστώ, είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Okay, Ευχαριστούμε κύριε Τζόνσον. Πολύ λεπτομερείς παρατηρήσεις σας. Κύριε Μπενιφέη, θέλετε να απαντήσετε. Φαντάζομαι πως θέλετε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την δουλειά που έχουμε κάνει μαζί, για τα καλά τους λόγια και ιδιαίτερος τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΕΡ. Θα ήθελα να του πω, να πω στον κύριο Τζόνσον, ότι αυτή η ανησυχία είναι κατανοητή. Θα ήταν όμως πολύ καλύτερο να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο. Θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες λεπτομέρειες σε μένα αλλά και στην Επιτροπή. Θα ήταν σαφέστατα πιο χρήσιμο πιο χρήσιμες για μένα, αλλά και στην Επιτροπή γενικότερα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς δίνεται στήριξη στην κοινωνία των πολιτών μέσω αυτής της γραμμή του προπολογισμού, την οποία ονομάσατε εισιτήριο εισόδου. Θα μπορούσατε να μου δώσετε λίγο περισσότερα νούμερα, προκειμένου να μπορέσω να επιχειρηματολογήσω αυτό το θέμα. Θα μπορούσατε να μου κάνετε μια αναλυτική κατανομή των ποσών και το πώς χρησιμοποιούνται. Συμφωνώ γενικά με τα όσα είπατε, μου φαίνονται πολύ λογικά. Θα ήθελα όμως να δω τις λεπτομέρειες μαζί σας. Okay, thank you. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ να καλωσορίσω ε, τους φιλοξενούμενους μας. Ένα από τα κρατήδια, τα πιο όμορφα κρατήδια της Γερμανίας είναι η κάτω Σαξονία. Και θέλω να ε, χαιρετήσω την Υπουργό Οικονομικών του κρατηδίου αυτού που είναι παρούσα σήμερα εδώ. Τροπολογίες μπορείτε να υποβάλλετε μέχρι τις 16 Ιουλίου, Δευτέρα. Τροπολογίες για τη γνωμοδότηση και για τον προϋπολογισμό. Και παρακαλώ μόνο στα αγγλικά. Ψηφοφορία πιθανότατα στην ΑΦΕΤ στις 29 Αυγούστου. Σημείο 7. Διάφορα. Έχετε κάποιο έτοιμα, όχι. Προσεχή συνεδρία 29 και 30 Αυγούστου. Κλείνω τη συνεδρίασή μας. Θα συνεχίσουμε ακριβώς στις 5 με το διευρυμένο Προεδρείο, μόνο δηλαδή συντονιστές και μέλη του Προεδρείου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα και να ευχαριστείτε το ποδόσφαιρο.